Good morning everyone. I think it's time to start our work. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ώρα νομίζω να ξεκινήσουμε τις σημερινές μας εργασίες με ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξη, δηλαδή μια μελέτη από την υπηρεσία EPRS ό,τι αφορά την ε, έκθεση για την εφαρμογή του 7ου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης, κοινή συζήτηση. Καταρχάς θα δώσω το λόγο στην κυρία Κατερίνα Καραμφίλοβα από το EPRS. Και έπειτα θα ακούσουμε την εισηγήτριά μας την κυρία Σέρμπου. Η κυρία Καραμφίλοβα. Uh, Καλημέρα σας. Είναι η τρίτη έκθεση που έχουμε ε, εκπονήσει για την Επιτροπή Ένβη, για την ε, της εφαρμογή. Πρώτα απ' όλα να σας παρουσιάσω αυτό το πρόγραμμα ως μέσο πολιτικής. Μετά θα σας παρουσιάσω τα βασικά μας ε, πορίσματα και θα ολοκληρώσω αναφέροντας ε, τις ε, πηγές, τα δεδομένα στα οποία βασιστήκαμε. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά το 7ο αυτό πρόγραμμα, εκεί βλέπουμε τους στόχους ε, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής μακροπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι το 2020 αλλά και πέραν του 2020. Ποιοι είναι οι στόχοι. Ο πρώτος στόχος είναι προτεραιότητες, παραδείγματος χάρη, προστασία, διατήρηση φυσικού κεφαλαίου. Ο δεύτερος στόχος ε, είναι ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές ε, και με ενεργειακή απόδοση και ο τρίτος στόχος είναι να μειωθούν ε, οι περιβαλλοντικές πιέσεις, ο κίνδυνος, η υγεία και την ευημερία. Αυτή είναι η βασική θεματική στόχη, όπως τους αποκαλώ εγώ, διότι συγκροτούν τις βασικές προτεραιότητες για τα κράτη-μέλη και καλύπτουν ουσιαστικά όλη την πολιτική περιβάλλοντος. Ποια είναι η λογική του προγράμματος. Πώς ε, θα επιτευχθούν αυτοί οι τρεις σταματικοί στόχοι, αν έχουμε βελτιωμένη εφαρμογή του στόχου 4, αν έχουμε περισσότερη γνώση και ε, στοιχεία για το στόχο 5, αν έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση για το στόχο 6 και αν έχουμε μια πιο συνεκτική πολιτική στο στόχο 7. Οι τέσσερις αυτοί στόχοι επόμενοι είναι το λεγόμενο enabling framework ε, που διευκολύνει δηλαδή την επίτευξη των στόχων. Α, τα βλέπετε και στην οθόνη. Ωραία, λοιπόν. Αυτοί οι 7 συνολικά στόχοι συμπληρώνονται και από δύο ειδικού στόχου, τον 8ο και τον 9ο που αντιμετωπίζουν τις ε, αστικές αλλά και λοιπές προκλήσεις του τομέα περιβάλλοντος και κλίματος. Οι λεγόμενοι οριζόντιοι στόχοι. Εννέα στόχοι λοιπόν συνολικά. Αυτή δεν είναι μόνο σε βυσπόθη, αλλά είναι δεσμευτικά, νομικά δεσμευτικό το πρόγραμμα και τα πρέπει τα θεσμικά όργανα της και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις κατάλληλες δράσεις. Υπάρχουν κάποιες πολιτικές, κάποιες δράσεις ε, που αναφέρονται και στο ίδιο το πρόγραμμα, αλλά με 10 λεπτά που έχω δεν να τα καλύψω όλα, ούτε και όλα τα πορίσματα, γι' αυτό θα σας παρουσιάσω μόνο την γενική εικόνα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος. Και έρχομαι λοιπόν με αυτά και με αυτά στο δεύτερο σημείο. Ποια είναι τα βασικά πορίσματα. Η εφαρμογή ε, για τους τρεις βασικούς θεματικούς στόχους, 1, 2, 3 και τους οριζόντιους στόχους, 8 και 9, αξιολογήθηκε με βάση αυτό που λέμε τις, ε, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης που είναι η συνεκτικότητα, η συνάφεια, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Προσθέσαμε σε αυτή τη δέσμη κριτηρίων ε, τη βάση γνώσεων που είναι ένα έκτο σημαντικό κριτήριο για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι η συνολική εικόνα εφαρμογής του προγράμματος. Τα πόρισματά μας είναι πρώτον οι τρεις βασικοί θεματικοί στόχοι, οι δύο οριζόντιοι στόχοι εξακολουθούν να είναι συναφείς και επίκαιρες ό,τι αφορά τις ανάγκες. Δεύτερο, υπάρχουν κάποια κενά στις γνώσεις μας σε ό,τι αφορά αυτούς τους βασικούς θεματικούς και οριζόντιους στόχους, αλλά και σε τομείς που δεν υπάρχει επαρκής αξιμοποίηση αυτής της ε, γνώσης που έχει συλλεγεί. Το τρίτο πόρισμα είναι ότι η συνεκτικότητα ε, είναι προβληματική, ιδίω ό,τι αφορά τον 1, 2 και 3, τους βασικούς θεματικού στόχους. Και η γεωργική πολιτική είναι το πιο σαφέ παράδειγμα. Και εδώ έχουμε ε, ένα πρόβλημα σε σχέση με του στόχου μα για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Τέταρτο πόρισμα, μεικτή η πρόοδος ό,τι αφορά την εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών, εξού και μεικτή η πρόοδος ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων. Η πιο προβληματική σε ό,τι αφορά την υλοποίηση τομής είναι η βιοπικιλότητα στο στόχο 1, η διαχείριση δεδομέ... συγγνώμη, αποβλήτων στο στόχο 2 και ποιότητα του αέρα και η χορύπανση στο στόχο 3. Για το 2020 δεν είναι και τόσο ελπιδοφόρα τα πράγματα, στη χειρότερη περίπτωση το στόχο 1, αλλά και στην καλύτερη περίπτωση είναι ασαφείς ε, οι προοπτικές για τον ε, στόχο 3, είναι δύσκολο να κάνουμε μια εκτίμηση. Δεν έχουμε παρκή στοιχεία στην παρούσα φάση. Πέμπτο πόρισμα, περιβαλλοντικές, κλιματικές πολιτικές. Είναι δαπανηρές, αλλά κατά ανάγκη δαπανηρές. Ωστόσο, δεν είναι παρκής ε, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών η χρηματοδότηση σε εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ επίσης έχουμε και ένα πρόβλημα με την ε, δαπάνη της χρηματοδότησης που υπάρχει. Βλέπουμε ότι δεν ε, υπάρχει παραπροβληματική εκτέλεση. Πάντως, παρά τα προβλήματα, υπάρχει προστέμενη αξία στο πρόγραμμα. Συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών μελών και της Ένωσης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα. Το 7ο πρόγραμμα θα μπορούσε να είναι μοντέλο για το επόμενο, το 8ο πρόγραμμα. Ωστόσο, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να απλουστευτεί, να υπάρξει μεγαλύτερη ε, καλύτερη επικοινωνία και πληροφόρηση σε εθνικό επίπεδο και να υπάρξει καλύτερη παρακολούθηση. Υπάρχουν στη μελέτη αρκετέ λεπτομέρειε για τον κάθε στόχο. Μπορείτε να δείτε πού βοηθάει αυτό το περιβάλλον που βοηθά αυτο το περιβαλλον ονόμασα enabling framework ή μπλοκάρει θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα για να διευκολύνω την ανάγνωση σας. σα ενδιαφέρει, για παράδειγμα, ο στόχος 1, που είναι η προστασία της διατήρησης διατήρηση της φύσης. Βλέπετε τι γίνεται με το στόχο 1, παραδείγματος χάρη, ε, τι γίνεται με την εφαρμογή. Έχουμε τα θέματα που αφορούν τη γνώση. Το δεύτερο ε, στόχο, μάλλον στον πρώτο στόχο, επίσης, έχουν τα θέματα χρηματοδότησης, και τα θέματα συνεκτικότητας. Το ίδιο ισχύει για τους άλλους στόχου, 2, 3, 8, 9. Επίσης μπορείτε να δείτε και κάποιες συστάσεις που στόχο είναι τη βελτίωση τη υλοποίηση σε κάθε στόχο. Δεν μπορούσαμε όμως να συνοψίσουμε τις συστάσεις μας, γιατί αυτό θα είχε νόημα μόνο στο συγκεκριμένο πλαίσιο της ε, συγκεκριμένη πολιτική. Μπορείτε λοιπόν να δείτε τις ε, συστάσεις αυτές μελετώντας ε, τα πορίσματά μας. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο και τελευταίο σημείο που είναι ποιε ήταν οι πηγές δεδομένων. Όπως ξέρετε πολλές είναι θέσιμες πληροφορίες για την υλοποίηση των μεμονωμένων ε, δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος. Δεν μπορέσαμε όμως τη μελέτη να καλύψουμε τα πάντα. Γιατί δεν θα είχαμε 300 σελίδες μόνος, αλλά χιλιάδες σελίδες και βέβαια δεν είναι αυτός ο στόχος μας ως ερευνητών. Αυτό που κάναμε αντίθετα ήταν να δούμε ακριβώς ε, τις ε, πηγές αυτές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να δίνουν στοιχεία για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προγράμματος. Και εδώ έχουμε δύο τέτοιες ε, πηγές στόχους. Η πρώτη είναι η έκθεση δικτών, Indicator Report που είχε δημοσιευθεί το Δεκέμβριο του 2016 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Σύντομα θα έχουμε την επικαιροποιημένη έκθεση και η δεύτερη είναι το Environmental Implementation Review που δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2017 και έχετε υιοθετήσει ψήφισμα αυτό το μήνα ε, σχετικά. Επίσης ζητήσαμε και από το ελεγκτικό συνέδριο να προετοιμάσει ε, την σύνοψη των βασικών τους ε, πορισμάτων για τις ειδικέ εκθέσεις περιβάλλοντος και κλιματικής πολιτικής. Αυτές οι τρεις πηγές μας δίνουν πολλές πληροφορίες και τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Δεν καλύπτουν όμως ε, οι πηγές αυτές και τους εννέα στόχους, το σύνολο δηλαδή του προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν και για να ξεπεράσουμε αυτή την πρόκληση, κάναμε μια διαβούλευση των εμπλεκομένων φορέων για να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα και συμπεριλάβαμε εδώ όλες τις δράσεις πολιτικής αυτό ευθυγραμμίζεται και με το πρόγραμμα που στο άρθρο 4 λέει ότι η εξελίξη του προγράμματο θα πρέπει μεταξύ άλλων να βασίζεται στι απόψει των ενδιαφερομένων φορέων. Πήραμε λοιπόν ε, τη συνεισφορά από ε, πολλούς, πολλά θεσμικά όργανα, από 22 κράτη-μέλη, διεθνείς οργανώσεις, ε, από οργανώσει που στηρίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και την προστασία της φύσης και από διάφορους ε, κλάδους της βιομηχανίας καθώς και ερευνητέ. Και βλέπετε ξεκάθαρα ποιες είναι οι απόψεις ε, των διαφόρων μπλεκομένων Στου ευρύτατου αυτούς τόμεις περιβάλλοντος κλιματική αλλαγής. Τα αποτελέσματα της διαβούλευση, από ό,τι ενημερώθηκα, θα σας βοηθήσουν και στο δικό σας έργο και γι' αυτό ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να διαβάσετε το παράρτημα 6. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνω, εκλογληρώνω αφού ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχαν στη διαβούλευση. Και επίσης να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Όργανο Περιβάλλοντος, το Αλληλεκτικό Συνέδριο που μας βοήθησαν στη λογική δεδομένων αλλά και του εξωτερικού μα έρευνε. θέλω να ευχαριστήσω από την Τεκνόπολη και την Τραϊνόμιξ. Είναι και εδώ εκπρόσωποι του αν θέλετε μπορείτε να τους θέσετε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ η PRS για τη μελέτη και τώρα. Η συγγήτρια, η κυρία Σάρμπο, έχει το λόγο. Καλημέρα σας. Συνάδελφε, πρόκειται για το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Είναι ευρύτερο πρόγραμμα, καλύπτει στόχους και νομοθετήματα. Αφορά ό,τι θέμα για το περιβάλλον μπορεί κανείς να φανταστεί. Και ήταν δύσκολη υπόθεση το να συντάξουμε αυτήν την έκθεση. Το EPRS ε, μας βοήθησε και ευχαριστούμε ιδίως την ε, Κατερίνα Και όπως είπαμε με τους εμπλεκόμενους συνοηθήκαμε και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, διάφορους φορείς, κράτη-μέλη μέσω των αντιπροσωπιών στις Βρυξέλλες, αλλά συνεργαστήκαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι αυτοί ανταποκρίθηκαν. Και επίσης συνεργαστήκαμε με την υπηρεσία περιβάλλοντος, το ελληνικό συνέδριο, τον οποίο η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Έπρεπε να είναι ευσύνοπτη αυτή η έκθεση, οπότε και δεν μπορέσαμε να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα. Γιατί βλέπετε ότι το σκηδοκειμένο είναι τα πιο σημαντικά, ό,τι θεωρήσαμε εμεί πιο σημαντικά τέλο πάντων. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα άξιζε να αναφερθούν. Και για αυτό το λόγο θα προτείνω κάποιε τροπολογίε, ούτω ώστε να καλύπτει περισσότερα πράγματα το κείμενο. Τώρα, οι παρατηρήσει για τα επιμένου ζητήματα περιέχονται στην έκθεση. Τώρα να μην ε, τα αναφέρουμε ένα-ένα, απλώς να σας κάνω μια σύνοψη από τα συμπεράσματα και συστάσεις. Νομίζω ότι η εικόνα είναι ανάμεικτη. Δηλαδή υπάρχουν κάποια θερεντικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και κάποια αρνητικά δηλαδή κάποια μέτωπα όπου η πρόοδος δεν ήταν ιδιαίτερα σημαντική σε μερικέ περιπτώσεις. Επίσης δεν έχω αρκετά στοιχεία για να κάνω μια πλήρη αξιολόγηση. Διάφορα ζητήματα ανέκυψαν όσον αφορά τη βελτίωση της υλοποίησης του προγράμματος. Πρώτα-πρώτα το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει κάποια συνοχή με τις άλλες πολιτικές ένωσες. Η αγροτική πολιτική επίσης τονίστηκε ότι πολλές φορές συγκρούεται με ε, το πρόγραμμα πλαίσιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό θίγει και τους τρεις στόχους. Το φυσικό κεφάλαιο, την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την αντιμετώπιση των κοινωνιών για την υγεία. Οπότε υπάρχει ιδίω γύρω στον αυτό το φυσικό κεφάλαιο αυξημένη πίεση ε, ας πούμε πρόβλημα είναι το ότι πετάμε το 1 τρίτο των παραγωμένων τροφίμων. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε και η αγροτική πολιτική να προσαρμοστεί. Να προσαρμοστεί στις προτεραιότητες του περιβάλλοντος. Να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες οικοσυστήματος και επίσης να μειώσουμε τα ιδιατροφής που πετάμε Οπότε θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια, όπως είπαμε, η συνεκτικότητα με την ε, αλληλευτική πολιτική, με τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Α, τώρα, να δούμε το θέμα των κενών στη γνώση. Έχουμε πολλά τέτοια κενά και σε σημαντικούς τομείς, όπως το συνδυασμένο αποτέλεσμα νανοηλικών και χημικών. Βέβαια έγινε κάποια πρόοδος πρόσφατα, αλλά, αλλά ακόμα υπάρχουν στοιχεία που καταδεικνύουν ότι στη χάραξη των πολιτικών δεν χρησιμοποιούμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες. Να, ας πούμε τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ή νομοθέτες δεν έχουν το θάρρος να εκμεταλλευτούν αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Βέβαια είναι και το θέμα της σύγκρουσης με άλλα συμφέροντα. Άρα η σε περιβάλλοντος θα πρέπει να βρει άλλους περισσότερους, καλύτερους δείκτες και έτσι να εποπτευθεί η υλοποίηση. Δεν θέλω να επικρίνω την υπηρεσία για το περιβάλλον. Το αντίθετο είναι πολύτιμα τα όσα συμπεράσματα και συστάσεις ε, προτείνει. Αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε όσον αφορά την υλοποίηση. Περισσότερους δείκτες, περισσότερα δεδομένα, ε, τα κρατή-μέλη, θα πρέπει να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης έχουμε θέμα πρόβλημα με την χρηματοδότηση σε επίπεδο κρατών μελών. Όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λείπουν τα χρήματα. Όμως, θα πρέπει να δούμε πώς τα δαπανούμε. Τα λέει το Ευρωπαϊκό Ελληνικό Συνέδριο. Πολλές φορές έχουμε διασπάθηση. Χαμένες ευκαιρίες. Ας πούμε, σε κάποιους τομείς που έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα, εκεί έχουμε πετύχει, ας πούμε, να βελτιώσουμε την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Μπορεί εδώ να κάνει πολλά Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσέξει περισσότερο, ούτως ώστε να πιάνουν τόπο οι κοινωνικοί φόροι. Θα πρέπει τώρα να δούμε πώς πάει η υλοποίηση του προγράμματος πλαισίου και πού μπορούμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις και συμφωνώ με τους άλλους εμπλεγόμενους που λένε ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει θετική επίδραση στην ε, πολιτική που ασκεί η Ένωση και αποκομίζουμε ωφέλη. Όμω υπάρχουν προβλήματα με την υλοποίηση, είναι θέμα συνεκτικότητα των πολιτικών, τα ένα στη γνώση και η χρηματοδότηση. Σε αυτούς τους τρει τομεί πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις. Μετά το 2020 είπαν περισσότεροι εμπλεκόμενοι, θέλουμε ένα άλλο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, οπότε το 8ο ας πούμε πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ευρύτερου ορίζοντες και συμφωνώ. Θα πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο πρόγραμμα πλαίσιο. Και να εκμεταλλευτούμε το τρέχον πρόγραμμα και κατόπιν των προβλημάτων υλοποίηση που εντοπίσαμε θα πρέπει κανείς να είναι επιφυλακτικός όσον αφορά αυτή τη διεύρυνση του ορίζοντα του πεδίου του μέλλοντος προγράμματος πλαισίου δεν τα πάμε τόσο καλά όσον αφορά την ε, επίτευξη των στόχων του 2020. Να δούμε τι θα κάνουμε με το φυσικό κεφάλαιο, την ποιότητα του αέρα και πάντως περιμένω να ακούσω τι σκέπτονται οι συνάδελφοι. Ακούσω τις προτάσεις, τις ιδέες τους. Όπως είπα, έπρεπε να είναι ευσύνοπτο το κείμενο και δεν μπόρεσα να καλύψω όσα ήθελα. Πάντως, θα προτείνω τροπολογίες και περιμένω πώς και πώς να ακούσω τη γνώμη σας. Ε, ευχαριστούμε κυρία Σάρμπου για την εισήγησή σας λέει η Πρόεδρος. Τώρα να στραφούμε προς τους σκιώδες εισηγητάς. Διάφορες πολιτικές ομάδες, πρώτο το ο κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εισηγήτρια για το πολύ καλό σχέδιο έκθεσης. Νομίζω πως περιέγραψε όλους τους σχετικούς τομείς. Συμφωνώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο το έργο της, το περιβάλλον βεβαίω. Έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Από την άλλη, οι στόχοι αυτοί πρέπει να καθοριστούν επακριβώς και πρώτα πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Εγώ θα συμφωνήσω με την αξιολόγηση των τριών στόχων προτεραιότητας. Κατά την αποψή μου η εφαρμογή δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώρες. Επίσης καμιά φορά υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Κάποιοι στόχοι εφαρμόζονται πάρα πολύ καλά, π.χ ο στόχος υπαριθμών 2, η οικονομία χαμηλό άνθρακα, αλλά πρέπει επίσης ε, να πούμε ότι αλλού η εφαρμογή είναι πολύ άσχημη. Να προσθέσω κάτι στην έκθεση. Πρώτα απ' όλα για τις βιώσιμες πόλεις και την ανάπτυξη τους. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για την προαστιοποίηση Η τεράστια οικισμή είναι μια πρόκληση για το μέλλον και θεωρώ ότι οι έννοιες αυτές ε, είναι ένα πρόβλημα η ανάπτυξη δηλαδή των πόλεων. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε το πώς αναπτύσσονται οι πόλεις και υπάρχουν και κάποια θέματα υγείας που σχετίζονται με αυτό και πρέπει να προσθεθούν στην έκθεση τώρα. Για την κοινή γεωργική πολιτική υπάρχουν κάποια κρίσιμα σημεία που τονίζει η αλλά επίσης πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και για τις δικές μας τις πολιτικές. Να αναφέρω, παραδείγματος χάρη, την στήριξη της πρώτης γενιάς βιοκαυσίμων σε κάποια κράτη-μέλη. Αυτό επηρεάζει την κοινή γεωργική πολιτική και επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. Πρέπει λοιπόν να επαναξιολογήσουμε με μια κριτική ματιά τις πολιτικές μας. Καμιά φορά υπάρχει και πρόβλημα με την αρχή της επικουρικότητας. Τα κρατημέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αρχή της επικουρικότητας, αλλά καμιά φορά ρίχνουμε όλο το βάρος στην επικουρικότητα και αυτό συγκρούεται με τους στόχους ε, της Ένωσης. Και πρέπει και αυτό να το αναφέρουμε στην έκθεση. Εγώ κάνα δύο τροπολογίες θα καταθέσω γιατί όπως είπα το σχέδιο έκθεσης είναι πάρα πολύ καλό. παρακολουθούμε και κάποια πράγματα που λέει η συγκήτρα. Εγώ συμφωνώ, πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής, να καθορίσουμε καλύτερα τους στόχους για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. έχει τον λόγο, ο κύριος με Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω εν μέρη με τον συνάδελφο. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή αρχή εδώ πέρα. Τα τελευταία τρία χρόνια που είμαι σε αυτήν την επιτροπή ασχολούμαι κυρίως με την κυκλική οικονομία την διαχείριση αποβλήτων, την φύση και την βιοπικιλότητα και βεβαίως στην Επιτροπή εμείς με τις εκπομπές και την ποιότητα του αέρα. Σε όλα αυτά λοιπόν έμαθα ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συχνά δεν εφαρμόζεται σωστά και αυτό επιβεβαιώθηκε σε κάποια έγγραφα αναφοράς, π.χ. την έκθεση ΣΟΥΡ 2015, την έκθεση για την κατάσταση της ε, φύσης και βεβαίως τα ακούσαμε και στην παρουσίαση όπου έχουμε την αξιολόγηση της εφαρμογής ε, της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής, αυτό το οποίο λέμε Environmental Implementation Review. Αν δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα στο σχέδιο, στο 7 σχέδιο δράση για το περιβάλλον, έχω αυτό το οποίο λέμε déjà vu, σαν να τα έχω ξαναδεί αυτά. Λέμε ότι χρειάζεται καλύτερη εφαρμογή, οπότε οτιδήποτε γράφουμε εμείς εδώ πέρα μένει στα χαρτιά. Δεν υπάρχουν δεδομένα, δεν υπάρχει γνώση υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, χρηματοδότησης κτλ. λοιπά. Τα προβλήματα λοιπόν είναι γνωστά, γνωρίζουμε από τι πάσχει ο ασθενής. Η έκθεση αυτή λοιπόν πρέπει να προχωρήσει παραπέρα από την γνωστή παράθεση των γνωστών προβλημάτων. Πρέπει να προτείνει λύσεις. Αυτό θα κάνω εγώ με τις τροπολογίες μου για να δώσουμε ένα μήνυμα Ακούσαμε και σήμερα το πρωί πάλι αυτές τις πληροφορίες από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Κοινοβουλίου. Οπότε, και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια και αναμένω βεβαίω την επικοδοκιμητική μας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Εκ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ την εισηγήτρια. Κάποια παράγματα αναφέρθηκαν, άλλοι στόχοι δεν θα επιτευχθούν τόσο γρήγορα, δεν υπάρχει πολιτική βούληση εντός του Κοινοβουλίου, αλλά δεν υπάρχει και εφαρμογή. Συμφωνώ και με την εισηγήτρια στην κριτική που ασκεί στην κοινή αγροτική πολιτική. Θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια για το φυσικό κεφάλαιο, όπως λέμε, όπως έχει δείξει η εξέταση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Βιοπικιλότητας. Φαίνεται ότι έχουν βλάβες τα οικοσυστήματα στην Ευρώπη βλέπουμε ότι δεν καταφέραμε να σταματήσουμε την εξαφάνιση των ειδών. 70% των προστατευόμενων ειδών εξακολουθούν να κινδυνεύουν. Εάν συνεχιστεί αυτή η καταστροφική τάση, τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Αν θέλουμε να την αναστρέψουμε, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα πάντα στην Ευρώπη. Γεωργία, συγκοινωνίες κτλ. Και να αναγνωρίσουμε πού είναι τα λάθη που οδηγούν σε μία μείωση της βιοπικιλότητας για να τα διορθώσουμε. Και βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε το τι γίνεται με την διαχείριση των λύκων στην κεντρική Ευρώπη. Ε, λένε κάποιοι ότι έχουν φτάσει σε ένα ανώτατο όριο λύκοι, και θα πρέπει να αρχίσουμε να τους πυροβολούμε. Πρέπει να ζούμε μαζί με τη φύση. Αυτά και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ. Thank you very much, Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση, κυρία Πρόεδρε, κυρία Συγήτρια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν τομείς που η κατάσταση διαφέρει. Είναι εντελώ διαφορετική. Ε, το λέμε, το ακούμε. Τελικά ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί κάποιοι τομείς να εξαφανιστούν. Η κατάσταση υποβαθμίζεται και υπάρχει υποχώρηση σε, σε περιπτώσεις όπως η βιοπικιλότητα για παράδειγμα. Όλα αυτά έχουν να μας πούν πολλά. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για τη φύση. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση σε αυτό το θέμα. Αν εστιάσουμε σε 5 και όχι 15 χρόνια ίσως πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις. Για την γλυφοσάτη ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ε, επικίνδυνο αυτό το ζανιοκτόνο. Η κατάσταση όμως ε, είναι τέτοια που θα έχουμε χειρότερες επιπτώσεις από την πριν. Τις αποφάσεις λοιπόν που λαμβάνουμε εδώ για το περιβάλλον θα πρέπει να τις ε, συσχετίζουμε με τις άλλες μας πολιτικές τα συζητάμε, είμαστε περήφανοι, ο ένας κοιτάει τον άλλον, η Κομισιόν εμάς, εμείς την Κομισιόν, χαιρόμαστε όλοι και τελικά γίνεται μια έκθεση, γίνεται μια έρευνα και βλέπουμε ότι δεν πάει τίποτα καλά. Ε, λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη όλα αυτά και να πούμε και στην Κομισιόν ότι εδώ έχουμε ευθύνε και τις ευθύνε αυτές πρέπει να τις αναλάβουμε. Τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει πρέπει να τις τηρήσουμε. Υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της Ένωσης. Μα γιατί. Φυσικά γιατί δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, δεν εφαρμόζουμε τις αποφάσεις μας. Επόμενο θέμα. Οι περιβαλλοντικές συμφωνίες, ε, κλίμα, ποσοστώσεις κτλ. Υπάρχουν ε, έρευνες και μελέτες που δείχνουν ότι ούτε εδώ η εφαρμογή είναι σωστή. Πρέπει να το ξαναπούμε πόσο σημαντική είναι η βιοπικιλότητα για το κλίμα. Μήπως η φύση θα έπρεπε να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της από μόνη της. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοια. Υπάρχει το ζήτημα επίσης των εκπομπών διοξιδιωτών του που έχει καταστροφικές συνέπειες για τη βιοπικιλότητα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια για το έργο της, πάρα πολύ σημαντικό. Όμως έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα αίτημα. Πρέπει η Επιτροπή να πάρει τα πράγματα, ε, την κατάσταση στα χέρια της. Και ο Επίτροπος Τίμπερμανς ε, πρέπει να καταλάβει δεν είναι small thing, δεν είναι μικρά πράγματα, όπως λέει αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί ο κ. Τίμπερμανς αυτά για τα οποία συζητάμε σήμερα. Αν δεν λάβουμε τις αποφάσεις από κοινού, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και αυτό είναι επικίνδυνο για τη φύση. Ευχαριστώ. Thank you uh, Ευχαριστώ. Εδώ κλείνω κατάλογο των σκιωδών και το λόγο έχουν άλλοι συνάδελφοι, άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Ποιος θέλει το λόγο, κύριος Λάινεν. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ το τμήμα μελετών για την μελέτη και την κυρία Σάμπο Ήμουν και εγώ της για την πολιτική μου ομάδα. Θυμάμαι την συνεργασία μας. Το έβδομο πρόγραμμα δράσης είναι καλό. Η εφαρμογή είναι μόνο μερικώς καλή, μπορούσε να είναι καλύτερη και ήδη υπόθηκε που είναι το πρόβλημα. Εμείς εδώ νομοθετούμε, συμφωνούν και 28, αλλά μετά δεν γίνεται τίποτα Σαν κράτη-μέλη και ήδη στο 7ο πρόγραμμα ε, είχαμε δώσει ειδικό βάρος στην εφαρμογή και αυτό κάνουμε και τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ενθαρρύνω την Κομισιόν να κάνει περισσότερα ως ε, θεματοφύλακας της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να δει ποιοι είναι οι λόγοι για την έλλειψη εφαρμογής και να μην ε, τραπεί αν δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία, να επιβάλλει κυρώσεις η διαδικασία επί παραβάση. Έχουμε δει ότι λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εγώ ζω σε μεθοριακή περιοχή και μπορώ να το επιβεβαιώσω ότι η πολιτική του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζεται και μόνο όταν υπάρξει απειλή διαδικασίας επί παραβάση εφαρμόζεται. Κάπου γίνονται τα πράγματα, κάπου αλλού. Όχι για την Natura 2000 και τις άλλες περιοχές προστασίας φύσης λείπουν λεφτά και θα πρέπει να υπάρξει μια, ένας μετασχηματισμός της οικονομίας μας ε, δεδομένη της προστασίας του κλίματος ε, και βλέπουμε ότι ε, δεν έχει υπάρξει αρκετό earmarking του προπολογισμού. Δηλαδή 80% των κονδυλίων δεν έχουν περιβαλλοντικούς όρους και μόνο 20% έχουν. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Υπάρχει βεβαίως τώρα πια και η Συμφωνία των Παρισίων ε, για την κλιματική προστασία και πρέπει να υπάρξει άρα μια μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής, ε, μια ένταξή της ε, Ήδη η αγροτική πολιτική έχει καθοριστεί ως ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί γιατί δεν σεβόμαστε ιδιαίτερως την φύση. Ένα πρόγραμμα θα πρέπει να έλθει οπωσδήποτε προσεχώς. Οι στόχοι βεβαίω εξακολουθούν να ισχύουν οι στόχοι του έβδομου. Δεν χρειάζεται να βρούμε νέα πράγματα, πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά τα οποία ήδη έχουμε, σε αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί και να φτιάξουμε ένα ωραίο πρόγραμμα. Ελπίζω η επόμενη Κομισιόν να επιδείξει περισσότερη έτσι, φιλοδοξία σε ζητήματα περιβάλλοντος από ότι η Επιτροπή Γιούνκερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μιλά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Βεβαίω η έκθεση αυτή βλέπει ως σοβαρό πρόβλημα την συνοχή της πολιτικής. Πράγματι θα πρέπει να πετύχουμε μια μεγάλη συνοχή της πολιτικής και αυτό σημαίνει να συμπληρώνονται τα αποτελέσματα, όχι το ένα να εξουδετερώνει το άλλο. Αν δούμε λοιπόν τα συμπεράσματα, έχω μια προσωπική παράκληση. Συνέπεια και συνοχή δεν μπορεί να σημαίνει ότι ο κάθε ένας ακολουθεί τη δική του κατεύθυνση. Πρέπει να έχουμε αυτούς τους κοινούς στόχους, η κοινή αγροτική πολιτική, έχει ως στόχο την επάρκεια τροφίμων. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να έχουμε αυτόν τον, να παραμελήσουμε αυτόν τον στόχο. Πρέπει λοιπόν να μετρήσουμε την κλιματική πολιτική για το εάν μπορεί να βοηθήσει να παράγουμε ποιοτικά και προσιτά τρόφιμα. Επίσης για το πρασίνισμα. Κοιτώντας τα μέτρα του πρασινίσματος βλέπουμε ότι 5% της καλλιεργήσιμης γης θα έπρεπε να έχει πάει στο πρασίνισμα. Και όμως οι γεωργοί το έκαναν στο 9%. Το πρόγραμμα αυτό λοιπόν υπάρχει ήδη εδώ και δύο χρόνια και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε ακόμα τις συνέπειες. Επίσης πρέπει να πούμε, αν την τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα η εισηγητρία, πρέπει να πούμε ότι έχουμε 300.000 εκτάρια εκτάσεις οικονομικής ε, οικολογικής ε, προτεραιότητας. Ε, αν σταματήσουμε εκεί πέρα να ψεκάσουμε, θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί βεβαίως ε, κάθε φορά που ραντίζουμε οργώνουμε και όλα στο χώμα και έτσι απελευθερώνεται διοξίδιο του άνθρακα. Επίσης, έχουμε την <coughs> επιβάρυνση μέσω της σπατάλης των τροφίμων 35% ε, της σπατάλης γίνεται στα νοικοκυριά. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να το δούμε, όχι μόνο να παραπεμε μόνο στην αγροτική πολιτική. Και αναφέρατε κάτι άλλο το οποίο ε, βεβαίως μου είναι πολύ αγαπητό, το καθαρό πόσιμο νερό που θέλουμε όλοι. Και αν δούμε το πόσιμο νερό, πρέπει να δούμε και τους σωλήνες, που είναι πολύ σάπιοι. Και η αποχέτευση επίσης πολύ σημαντική και πρέπει να τονιστεί και κάτι ακόμα για τη γεωργία. Θεωρώ ότι η γεωργία ε, έχει συμφέρον να βλάψει τη φύση. Οι γεωργοί ζουν από αυτό και θέλουν να τα δώσουν στην επόμενη γενιά. Και αυτό πρέπει νομίζω σε μια τέτοια έκθεση να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θέλει άλλο το λόγο. If not, I turn to the Commission. Uh, I have Mr. Rosenstock. Θα σας τροφούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, κύριε. Κύριε Ρόζεν Στοκ. Thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την τόσο αξιόλογη έκθεση. Πάρα πολύ ευχαριστώ το ότι επιβεβαιώνεται από την έκθεση ότι είναι χρήσιμο εργαλείο το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο τόσο ώστε να πιάσουν τόπο οι πολιτικέ μα. Πολύ πολύ θετικά τα συμπεράσματα της κυρίας Σάρμπου. Επίση ε, το, το, το timing ήταν πάρα πολύ εύστοχο όσον αφορά αυτή την έκθεση γιατί τώρα μπορούμε πλήρω να ε, λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματά σας ε, για τη διαδικασία της αξιολόγησης που μόλις ξεκίνησε και έχουμε δημοσιοποιήσει αρχές Νοεμβρίου το σχετικό χάρτη πορείας ο εκεί προβλέπεται η μεθοδολογία της αξιολόγησης μπορείτε όλα αυτά να τα βρείτε στο website της Κομισιόν Better Regulation επίσης είναι πολύ θετική η προσέγγιση για την αξιολόγηση της εισηγήτριας όλα αυτά που λέει συμπληρώνει αυτά τα οποία εμείς έχουμε σκεφτεί για τις προτεραιότητες του προγράμματος, για, τις, ε, ε, για το, το, το ρόλο των υπηρεσιών περιβάλλοντος, στρατηγικός ρόλος, ε, η δομή του προγράμματος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε το αν έχουμε τη σωστή στρατηγική για το περιβάλλον. Και εάν έτσι έχουμε πιο πολύ προβληψιμότητα ε, από πλευράς κρατών μελών και από πλευράς δικής μας, αν υπάρχουν οι συνέργειες, αν προσφέρονται έτσι κάποιες ευκαιρίες και αν υπάρχει έτσι και οικονομία στην χρήση των πόρων, οπότε ακριβώς να προχωρήσουμε στην υλοποίηση που εσείς αναφερθήκατε να καλύψουν τα προβλήματα της χρηματοδότησης, των κενών στη γνώση, της εφαρμογής τελικά. Όπως είπε κάποιος από αυτούς που έλαβαν το λόγο τώρα στο τέλος. Επίσης, για τη διαδικασία της επιλογής των δικτών, να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες 1 έως 3, ό,τι προτείνει δηλαδή η υπηρεσία περιβάλλοντος, αλλά αν ληφθεί υπόψη και υπόθεση της διακυβέρνησης, ή διαβουλεύσεις, να έχουμε πιο στοχευμένες διαβουλεύσεις. Το καλοκαίρι του 18 θα έχει η αξιολόγησή μας και εν να σχολιάσω τις τέσσερις ε, συστάσεις σας. Πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες που προβλέπει η Επιτροπή για αρχάς του 2018 θα αντιστοιχούν σε αυτά που σας απασχολούν. Για παράδειγμα, για το νερό, για τα πλαστικά και για μια βιώσιμη στρατηγική χρηματοδότηση. Όλα αυτά θα κρυφθούν τις προτάσεις μας αρχάς του 2018. Πριν το τέλος του 2017 επίσης θα υπάρξει μια ανακοίνωση για κάποιες επιλογές εξυγχρονισμού της ε, ΚΑΠ, τα είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, αυτή η μεταρρύθμιση θα μεγιστοποιήσει τη συμβολή της ΚΑΠ όσον αφορά τις ε, πρωτοβουλίες μας, τη Συμφωνία των Παρισίων, τους διώσιμους στόχους κλπ. Τα είπατε κι εσείς. Οι πιο σημαντικές προκλήσεις για τον χρόνο ε, βέβαια θα είναι το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Τον Μάιο θα διατυπώσουμε τη σχετική πρόταση εποπτεία, διαφάνεια, λογοδοσία, όλα αυτά θα είναι σημεία σημαντικά. Επίσης, θα οι δαπάνες για το περιβάλλον από τον προϋπολογισμό και αυτό το θίξατε. Καλύτερα πολλά ταμεία και πόρους. Έχουμε το live, αλλά και σε άλλα ταμεία προβλέπεται χρηματοδότηση για το περιβάλλον ιδίως σε διοπτικά ταμεία, συνοχής. Είπαμε να αρθούν αυτά τα κοινά στη γνώση και συνεχίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε τη σχετική κοινότητα για τη γνώση του περιβάλλοντος. Αυτό θα καλύψει. Και θα έχουμε αρχάς του 18 την έγκριση του προγράμματος εποπτείας για τους στρατηγικούς στόχους και έτσι προχωράμε στην αξιολόγηση. Άρα η συνοχή θα είναι το πιο σημαντικό. Ε, ευχαριστούμε. Και σας που θέλετε να δευτερολογήσετε, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Μάλιστα, λέει η συγγήτρια. Και σας ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τις ιδέες σας, για τις απόψεις σας και την Επιτροπή να ευχαριστήσω. Και συμφωνώ 100%. ότι με τις τροπολογίες θα εντυπώσουμε τις προτάσεις μας τις λύσεις για τις πόλεις, μεταφορές, τον, την ατμόσφαιρα, διατροφική ασφάλεια. Όπως τα είπατε, είναι πολύ σημαντικό για τα τρόφιμα που πετάμε. Περιμένω προτάσεις από εσά. Μαζί, μαζί θα ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή. Και αυτό θα είναι το σωστό μήνυμα που θα στείλει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Και πάλι ευχαριστώ. Περιμένω τις τροπολογίες σας. Ε, εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε όσους κάνουν τη μελέτη την συγκίτρια, όσους λαμβάνουν στη συζήτηση και σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία είναι 5 Δεκεμβρίου για τις τροπολογίες. 11 ώρα το πρωί θα ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ στις 27 Δευτέρα του χρόνου. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση. In half an hour. Ten, um, half past ten. Ψηφοφορία στις 10.30. Μέχρι τότε διαλυματάκι. Hello everyone. Maybe you would like to take your seats. Σας ευχαριστώ παρακαλώ καθίστε. So we can start the voting procedure because we still have work. Ξεκινήσουμε την ψηφοφορία γιατί έχουμε και δουλειές μετά. ξεκινήσουμε κάποιες ε, ψηφοφορίες γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, για να δούμε κάθε είστε όλοι βλέπω. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία σήμερα. Έχουμε την ε, αντίρρηση για τα φωσφορούχα στο κρέας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχουμε γλυκαντικά σε προϊόντα φούρνου, άρχιτη ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται. ψηφίζουμε τώρα τεχνικές προδιαγραφές για ένα σύστημα εχνηλασιμότητας για καπνικά προϊόντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται. Ξανά. Τεχνικές προδιαγραφές για χαρακτηριστικά ασφαλείας για καπνικά προϊόντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε. Ενεργός ουσία γλυφοσάτη. Περί ανανέωσης της έγκρισης. Άρχεται η ψηφοφορία. και απορρίπτεται. Το επόμενο είναι μια παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών καλλιντικών σε ζώα. Προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία απόφαση του Συμβουλίου για την σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Ένωσης για την σύνδεση των συστημάτων εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Άλλη μια προφορική ερώτηση. Επανερχόμαστε στην απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για τη δημιουργία καλλιτικών, γιατί αφορά και το Συμβούλιο. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία ξανά. Παγκόσμια απαγόρευση δοκιμών σε ζώα για τα καλλιτικά. Τώρα είναι ε, προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο. Πέρας και εγκρίνεται. Τώρα περνάμε σε πιο δύσκολα θέματα. Διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών, θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης 20.030, Εισηγητή ο κύριος Φαρία. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές συμβαστική 2 υπέρ ευχαριστώ εγκρίνεται 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75, όχι, 86 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90, όχι. 91 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλίας 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αλίας 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται.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 απορρίπτεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, ελέγχουμε την 111, ελέγχουμε την 111, άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε, νομίζω, ναι απορρίφθηκε. 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αλία 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ελέγχουμε. Την 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίφθηκε. 126. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130, όχι, 131 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 5 αλίας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 της αλίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά ποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά ποχές δεν είδα τι κάνανε οι σοσιαλιστές. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 16 αλίας. Τι θέλετε να ελέγξουμε, την 140, εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. And is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε. Ευχαριστώ. Άλλαξαν οι ψηφοφορίε, οι πλειοψηφίε εδώ και μπερδεύτηκα. Πηγαίνουμε σε συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 149 και 153 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 151 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Τώρα τι ψηφίζουμε. Την τροπολογία 95 υπέρ αν απορριφθεί η συμβιβαστική, ψηφίζουμε αυτές που κάλυπτε. Και αυτό κάνουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τροπολογία 95. Ψήφι υπέρ. Μα απορρίφθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε τη συμβαστική 8, να την ελέγξουμε. Compromise 8. Συμβιβαστική 8. Δεν ψηφίζετε. Καλά. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Άρα ψηφίζουμε τις τροπολογίες. Και ξεκινάμε ξανά. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 183. Έχει αρχίσει η ψηφοφορία, πέρας τώρα, εγκρίνεται.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 εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 182 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 191 και αλληλεία» 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τραν 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογίες 201-202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 209 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 210 έχουμε χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές 211 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.16 υπέρ κατά αποχές ποιος είναι υπέρ του 2.16 κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Χωριστή ψηφοφορία στο 24 μέρος πρώτο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, μέρος δεύτερο υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική έννοια υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 11 υπέρ κατά αποχές ποιος είναι υπέρ τραν 11 κατά αποχές εγκρίνεται 2.40 υπέρ Να δούμε λοιπόν. Τραν 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ECR θα ψηφίσει. Το έτσι, από περίεργεια ρωτάω. Λοιπόν, πέρασε. Εγκρίνεται. 2.40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.44 υπέρ κατά αποχές ε, δεν σηκώνετε χεράκια 2.44 υπέρ κατά απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.46 υπέρ κατά αποχές να επαληθευτεί και πέρας εγκρίνεται 2.47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ 53 κατά αποχές εγκρίνεται 2.54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.57 χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 261 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 262 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 263 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 264 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 265 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3,10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική αναφορά 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάντα τραν, συνεχίζουμε, όχι, όχι, τελείωσε, μάλιστα, ωραία. Τώρα οι δικές μας τροπολογίες, 22 υπέρ, 1 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 και σαν αιτιολογική αναφορά 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ όχι 5 εγκρίθηκε άρα αυτή καταπίπτει. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κραν ιδεολογική αναφορά 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 και τραν τη αναφορά 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 και τραν 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 και τραν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 και 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 και 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν τη λογική αναφορά 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές ποιος είναι υπέρ 48 κατά να την επαληθεύσουμε λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας και απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτονται. 50 υπέρ κατά ποιοι είναι υπέρ 50 εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 52 ψηφίζουμε Ίσως προχωρούμε πολύ γρήγορα. Δεν προφταίνει να σηκώσετε τα χέρια σας. Πέρα στις και απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά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 Αλίας 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αλίας 8 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Τώρα έχουμε μία σειρά τροπολογιών από την Επιτροπή Αλίας Απλώ θα πω τα ονόματα. Δέκατα μάλλον τον αριθμό της τροπολογίας. 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Α, για να ξαναδούμε, ξανασηκώστε τα χέρια για το 15 υπέρ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 Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Α, αποχές 24 υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 30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 Κατά. Ξανασηκώστε τα χέρια σας για το 42. Υπέρ. Κατά. Ποχές. Ας γίνει λειτουργός έλεγχος για το 42. Πέρας. Ναι, με σαφή διαφορά. Εγκρίνεται 43. Υπέρ. Κατά. Α, αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Και εγκρίνεται. Η επόμενη ψηφοφορία αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αρχίζουμε. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 6α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 6β. Υπέρ. Να κάνουμε έλεγχο για το 6α. Ναι, συμβαστική είναι. 6α. Ψηφίζουμε. And closed. Rejected και απορρίπτεται. Για το 6β συμβαστική. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, ανάποδα, ανάποδα. 6β. Ψηφίζομαι. Δεν ψηφίσατε όλοι. Καλά, όποιος θέλει. Πέρασε. Adopted. 77. 77. Α, την καλύπτει. Η 6. Α, β. Καλά. 12 υπέρ. Κατά. Αποχέ. 79 υπέρ. Συμβαστική 5α υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 5β Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς. Το ίδιο, το ίδιο θα είναι. 5α ψηφίζομαι. And is close. Πέρος. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5 β υπέρ. Σχεδόν κανένα δεν σηκώνει το χέρι του. 5 β υπέρ κατά ας γίνει έλεγχος επαλήθευσης και ψηφίζομαι για το 5 β πέρας και σε αυτή την περίπτωση έχουμε απόρριψη 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 έλεγχος το προτείνετε. Ζητείτε επαλήθευση ηλεκτρονική. Μάλιστα. Ψηφίζουμε για το 13. Πέρασε. Και απορρίπτω. 80. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά. Abstentions. Αποχές. Απ' την άλλη δεν βλέπω χέρι, οπότε επανάληψη. 4 υπέρ κατά. Επαλήθευση. Ψηφίζομαι. Μα τι γίνεται, άλλα ψηφίζεται σε κάθε συμβαστική, τέλος πάντων. Εγκρίνεται. 84. Πώς? Okay, so 87. 87, who is in favor? 87. Υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. 88. Υπέρ, κατά, αποχές, 89. Υπέρ, κατά, αποχές, 90. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται, διορθώνει η πρώτη. 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 Θέλετε ηλεκτρονική Καλός Καλώς ψηφίζουμε για το 18. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται. 101 in favor. Against. 101. Υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Χωριστή ψηφορία για το 102. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτωται. Ή όχι επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα γιατί πολλοί από σας απέσχουν 102 δεύτερο τμήμα. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Α, αποχές. Απορρίπτεται. 104 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά Α, αποχές. Επαλήθευση για το 106. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά. Αποχές. 3, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 109, υπέρ κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά Α, απορρίπτεται 23 υπέρ κατά Αποχέ. επαλήθευση για το 23 ψηφίζουμε πέρασε εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 114 εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Στο 117 είναι κανείς κατά της προφορικής. Οπότε θα ψηφιστεί ομού. Με την 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Το ίδιο ισχύει και στο 118. Ένσταση για την προφορική. Όχι. Ψηφίζουμε και τις δύο. 118 με την ε, προφορική της τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το ίδιο και για το 119 δεν υπάρχει ένσταση. Ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε με την προφορική υπερκαταποχή. Εγκρίνεται. Το ίδιο για το 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πηγαίνουμε στην 121 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτει, 124 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές. Ελέγχουμε την 29, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται.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 Πού πάμε, πού πάμε. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. And close. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά 75 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το σύνολο της τροποποίησης και της άρχεται η ψηφοφορία. and it is adopted. Εγκρίθηκε. Επόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η συμβιβαστική πρόταση για το ETS. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Αυτά ήταν. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας ε, στις ψηφοφορίες. Ah, right in time. Αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας. Πρώτο θέμα, πρόταση ψηφίσματος για την κατάργηση σε παγκόσμιο επίπεδο των δοκιμών σε ζώα για τη δημιουργία καλλιτικών προϊόντων. Έχουμε μια σειρά από συνεισηγητές αν δεν εκπροσωπεί κάποιος την κυρία Πιέτη θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που βάλατε αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τους πολίτες της Ένωσης. Και γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα και ε, υπάρχει και μεγάλη ανταλλαγή πληροφοριών. Θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε την ηγετική της θέση και στάση και έδειξε στον ε, υπόλοιπο κόσμο ότι μπορούμε να είμαστε σε μια κατάσταση όπου τα καλλιντικά προϊόντα δεν θα δημιουργούνται μετά από δοκιμές σε ζώα. Και γιατί το αναφέρω αυτό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα πλήρη, ε, μια πλήρη απαγόρευση στις δοκιμές σε ζώα, καθώς και παγκόσμια απαγόρευση στην θέση στο εμπόριο καλλιτικών που ε, έχουν δοκιμαστεί σε ζώα. Και βέβαια από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ αυτή η απαγόρευση έχουμε θετικά αποτελέσματα. Τα βλέπουμε. Πιστεύουμε ότι και για τη βιομηχανία ήταν θετικά τα αποτελέσματα, γιατί υπήρχαν φόβοι ότι θα πληγεί η βιομηχανία λόγω αυτής της απαγόρευσης. Βλέπουμε όμως πως ανθεί η βιομηχανία γιατί πλέον ε, βασίζεται στην καινοτομία. Επίσης ε, γίνεται πολλή έρευνα σε αναλλακτικέ μεθόδους δοκιμών. Και αυτό επίσης έφτωσε θετικά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να πούμε πως ε, η σύγχρονη επιστήμη δράζεται σε καινοτόμες τεχνολογίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα. Το μήνυμά μου το βασικό αυτό είναι για σήμερα και πιστεύω ότι χάρη στην δική μας πρωτοβουλία θέλουμε το μήνυμα αυτό να το περάσουμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πιστεύω ότι πρέπει να υποστηριχθεί η δράση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Και ελπίζω να στηρίξουν ε, τα θεσμικά αυτά όργανα και τις δικές μας δράσεις. Θα ζητούμε λοιπόν ε, να προωθήσουν την παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα για την δημιουργία καλλιντικών. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω. Όταν μιλάμε για αναλλακτικέ μεθόδου δοκιμών, αντί δηλαδή δοκιμών σε ζώα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αυτές οι εναλλακτικέ μέθοδοι να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Ούτε θέλουμε βέβαια και να παρακολύσουμε την καινοτομία. Αυτά που λέμε είναι ότι υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι, έχουν εγκριθεί, είναι καλές και δείχνουν ότι εφόσον υπάρχει ε, παγκόσμια απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να έχουμε ποιοτικά καλλιντικά. Και πιο ποιοτικά, θα έλεγα, καλλιντικά ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, έχει περάσει αυτό το μήνυμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Βλέπουμε ότι η σταδιακή κατάργηση των δοκιμών σε ζώα είναι εφικτή και μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Εξού, λοιπόν, και καταθέσαμε αυτή την πρωτοβουλία. Στόχος μας είναι αυτή η παγκόσμια παγόρευση να εγκριθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ με οτιδήποτε είπε η Μίριαμ. Και έχουμε βεβαίω και τα όσα γίνονται στη Νέα Ζηλανδία, του Γουατεμάλα, σε διαφορετικέ χώρε. όπου έχουμε βεβαίω διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν θα μιλήσω εγώ για απαγορεύσει και το τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα θέλουμε να απαγορεύσουμε πράγματα και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και είναι βεβαίω κάτι διπλωματικό πάμε, στον ΟΗΕ για αυτό το θέμα, να ενθαρρύνουμε τον ΟΗΕ να εμπλακεί και τα μέλη του. Οπότε, με βάση αυτά θα ήθελα να πω το εξής. Ότι δηλαδή η Επιτροπή μας υιοθετεί την διατύπωση όπως προτείνεται από ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτών από διάφορες πολιτικές ομάδες και να μην ε, προσθέσουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καμιά φορά αυτό είναι σωστό βεβαίω να μιλάμε εντάξει, μεταξύ μα ή στην Κομισιόν, αλλά πρέπει να είμαστε εστιασμένοι. Έχετε ουσιαστικά σημεία. Δεν είναι τώρα εδώ πέρα το σημείο να προσθέσουμε οτιδήποτε μας ενδιαφέρει για την ευζοία των ζώων λίγα λόγια και σωστά για να έχουμε και υποστήριξη από το 80% των χωρών που δεν ακολουθούν αυτή την πολιτική. Σας ευχαριστώ λοιπόν και ελπίζω να μπορέσουν να το υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ Κύριε Ρής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, φυσικά και συμφωνώ με όλα όσα ακούσαμε. Και βέβαια έδειξε το δρόμο η ψηφοφορία προηγουμένω. Είδαμε πόσο ευρία είναι η πλειοψηφία υπέρ του σχετικού ψηφίσματος. Ε, να σας πω τώρα ε, ένα-δύο πραγματάκια ε, εδώ και πέντε χρόνια έχει τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά αυτή την γενική απαγόρευση των δοκιμών στα ζώα. Και έχουμε βέβαια 115 εκατομμύρια ζώα τα οποία θυσιάζονται στα εργαστήρια 200 χρόνων παγκοσμίω. Παγκοσμίω το χρόνο. Α, υπάρχει βέβαια μια πίεση από πλευρά του κόσμου. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει έχουν κινητοποιηθεί και οι καταναλωτέ. Όλο ένα και περισσότερο. Είναι όλο ένα και πιο σαφέ ότι προτιμούν τα προϊόντα που λένε ότι δεν έχουν περάσει από τέτοιε εργαστηριακέ δοκιμές επί Ο κόσμος έχει ευαισθησία για το πόσο υποφέρουν ε, τα Οπότε είπαμε τελικά είναι τέσσερις στις πέντε χώρες που δεν έχουν απαγορεύσει. Ισραήλ, Ινδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία. Βλέπουμε ότι οι χώρες σιγά σιγά αρχίζουν και μετακινούνται. Πάνε προς αυτήν την απαγόρευση και σύντομα θα το κάνει η Νότια Κορέα, η Αυστραλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ήδη ήταν η πρώτη που ε, έχει περάσει τέτοια ψηφίσματα και είπαμε ότι πέντε χρόνια μετά την απόφαση της γενικής απαγόρευσης ε, παραμένει πρώτη βιομηχανία στην Ευρώπη. Μιλούμε για δύο εκατομμύρια θέσεων εργασίας. Μιλούμε για επενδύσεις εκατομμυρίων ετησίως για να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να μην γίνονται αυτές οι δοκιμές. Συνεργασία, ε, προγράμματα, ε, διάφορους σπόνσορες την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως. Οπότε θα πρέπει ο κλάδος να συνεχίσει αυτή την συνεργασία και μακροπρόθεσμα να συνεχιστεί η αναζήτηση εναλλακτικών. Και, α, και ένα άλλο πραγματάκι. Θέλω κάτι να αλλάξει στο κοινό κείμενο. Κάτι να προσθέσω. Ε, ε, αυτή την έρευνα για εναλλακτικέ την χρηματοδοτεί ε, ο κλάδος. θα έπρεπε να συμβάλλουν σε αυτή την εναλλακτική έρευνα και τα πανεπιστήμια να προωθεί αυτό το ψήφισμα γιατί υπάρχει ευρύτατη συνένεση στην Επιτροπή μας αλλά και στο Κοινοβούλιο γενικότερα. ΕΚ. Κύρια Πρόεδρε, ευχαριστώ που συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα μια παγκόσμια απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα για καλλιτικά. Έχει αργήσει όλας. Ήδη και σήμερα έχουμε τέτοια προϊόντα και βεβαίως δεν υπάρχει ζήτημα ανθρώπινης ασφαλείας. Επιπλέον έχουμε μέσω του συνδυασμού των υφιστάμενων δραστικών ουσιών να έχουμε νέα προϊόντα χωρίς να χρειάζονται νέα πειράματα σε ζώα. Παρά λοιπόν τις εναλλακτικέ υπάρχουν εκατομμύρια τέτοια πειράματα κάθε χρόνια για να βγάλουμε μια νέα κρέμα κατά των ρητίδων. Δηλαδή πόσο άθλιος πρέπει να είναι κανείς για να κάνει κάτι τέτοιο. Σε πολλές ε, τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, βεβαίως βλέπουμε ότι αυτά τα προωθεί η βιομηχανία γιατί δεν θέλει να κάνει κάτι χωρίς πειράματα σε ζώα. Θα πρέπει λοιπόν να τους οθήσουμε προς την σωστή κατεύθυνση και να πω κάτι το εξής. Ναι, εντάξει, ακούμε, να ακούσουμε τις επιθυμίες των εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης ε, που είναι υπέρ μιας τέτοιας απαγόρευσης. Και θα είμαστε στην σωστή κατεύθυνση στο σωστό δρόμο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Εδώ πέρα κλείνει ο καταλόγος των μιλτών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος για να δω. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμπαθάτε με που άργησα. Ήμουν στην Επιτροπή Αναφορών Έχω και εγώ προσυπογράψει αυτό το ψήφισμα. Χαίρομαι που συμμετέσχουν. Αλλά δεν άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι. Πάντως να σας τονίσω το εξή. Είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ευρώπη και το Κοινοβούλιο στη διεθνή σκηνή, στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις να προωθήσουν την υπόθεση αυτή της απαγόρευσης για τα καλλιντικά της απαγόρευσης των δοκιμών. Υπάρχουν πολλά παραθυράκια και κενά στην νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρξει αυθεντική, ουσιαστική απαγόρευση των δοκιμών στα ζώα για τα καλλιντικά. Αυτό θα ζητήσουμε να υπάρξει περιορισμός, απαγόρευση διεθνώς. Για το Stop Vivisection υπέγραψαν την πρωτοβουλία 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι και όλοι οι κλάδοι. La sperimentazione eh, sugli animali. Ehm, Για αυτή την ζωοτομή, τέλος πάντων, στα ζώα. Οπότε θα πρέπει για κάθε κλάδο και τομέα να σταματήσουν τα τεστ στα ζώα και αυτό για την καλομεταχείριση των ζώων να ισχύσει διεθνώς γιατί εδώ παίζεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη μέσα διάταξη είναι η παραβίαση σχετικής νομοθεσίας εις βάρος των ζώων. Έχουμε, ξέρετε, πάρα πολλές αναφορές από πολίτες στην Ευρώπη. Έτσι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Δεν θα πρέπει να αδρανούν άλλο τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστούμε η κυρία Γκροστέτ. Πολύ καιρό είμαι βουλευτής και θυμάμαι συζητήσεις πώς να πάρα πολύ έντονες, φορτισμένες όσον αφορά την υπόθεση αυτή για τη ε, τεστ και τις δοκιμές στα Και σήμερα απαγορεύονται αυτού του είδους οι δοκιμές. Ε, τελικά κατέβαλε πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες ε, ο κλάδος για να βρει εναλλακτικέ. Είναι σημαντικό αυτή η απαγόρευση να ισχύσει παντού να προβάλλει τη θέση της Ευρωπαϊκής, να ακουστεί η φωνή της. Να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια καινοτομία στον κλάδο των καλλιντικών. Είναι κάτι το καλό. Είναι σημαντικό να το τονίζουμε και είναι σημαντικό να είναι παγκόσμια γενική η απαγόρευση. Μα είναι και θέμα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας μας. Όντως, κοστίζει η αναζήτηση και επεξεργασία και ανάπτυξη των εναλλακτικών. Αλλά τα κατάφερε ευτυχώς η βιομηχανία. Ήταν αναγκαία αυτή η απαγόρευση. Και γι' αυτό χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια. Τώρα, α, σε σχέση με την προλαλή σας, συνάδελφο, έχω να πω το εξή. Προσοχή. Συμφωνούμε όλοι για την απαγόρευση όσον αφορά τα καλλιντικά και συμφωνούμε εδώ και πολύ καιρό. Όμως, Προσοχή, προσοχή λίγο. Γιατί δεν θέλουμε να υπάρξει το ίδιο όσον αφορά την επιστημονική και την ιατρική έρευνα. Γιατί υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, έστω και σπάνιες, αλλά πολύ σημαντικές για την ιατρική, όπου δυστυχώς ακόμα χρειάζονται να γίνονται δοκιμές επί των ζώων. Οπότε, ναι, ναι, να προσέξουμε την καλομεταχείριση των ζώων. Όμως ακόμη υπάρχουν τομεί έρευνα στα πλαίσια της ιατρικής όπου δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τα τεστ τα ζώα. Προσοχή επομένως σε λίγα χρόνια ίσως μακάρι να τα καταφέρουμε να είναι εφικτό κάτι τέτοιο αλλά τώρα να μην επεκταθεί η απαγόρευση στην ιατρική έρευνα. Ευχαριστούμε, λέει η πρόεδρος και δίνει το λόγο στην κυρία Ντορνανό. Η καταπολέμηση και η απαγόρευση μας βρίσκει σύμφωνος. Συμφωνούμε με αυτό το κείμενο. Αποφάσισε η Επιτροπή μας να απασχοληθεί με το θέμα και ανέκαθεν εγώ έλεγα ναι σε αυτό. Και συντονίστρια είπα θα πρέπει να γίνει η γενική απαγόρευση όχι μόνο για τα καλλιντικά αλλά ε, με την ε, απαγόρευση οδηγηθήκαμε σε αναζήτηση εναλλακτικών και πέραν των καλλιντικών, αλλά θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα της ε, βιομηχανίας των καλλιντικών. Τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια που χρησιμοποιούνται ε, και για τρόφιμα και για απορριπαντικά και για φάρμακα. Υπάρχει επομένως ένα νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν στα πλαίσια της νομοθεσίας του ΡΙΤΣ εξαιρέσεις που επιτρέπουν. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσον θα διευρυνθεί η απαγόρευση, θα περιταθεί στα πάντα. Θα πρέπει, ναι, να απαγορεύσουμε για τα καλλιντικά. Αλλά αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνο. Άπαξ και η θέση σε εμπορία των προϊόντων που έχουν περάσει από τέτοιε δοκιμέ γίνεται εκτό. Το Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Το 2 Ιούλιο είχαμε μια συγκεκριμένη μάρκα που είχε τοποθετηθεί κατά αυτών των δοκιμών και υπέκυψε όμως τελικά από κάποια ασυργή αγορά και τελικά επέτρεψε να γίνονται δοκιμές σε εκείνη τη χώρα επί των ζώων. Ε, για αυτό και συμφωνώ στα πλαίσια του ΟΗΕ να γίνει διεθνής συνθήκη και να απαγορεύει αυτές τις δοκιμές που αποσκοπούν στην κατασκευή καλλιτικών και όχι μόνο. Και ευχαριστώ. Ε, εμείς ευχαριστούμε. Άλλος θέλει το λόγο. Όχι, λέει ο Πρόεδρος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κάτι. Or not. Ε, όχι, δεν ξέρω. Μάλλον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τη σημερινή συζήτηση, η οποία πράγματι ε, συνεισφέρει στο θέμα αυτό της απαγόρευσης των δοκιμών σε ζώα ε, για τα καλλιντικά. Πολλές φορές έχουμε πει πόση σημασία αποδίδουμε ως Κομισιόν στο θέμα <coughs> και Μάλιστα υπευλήθη πρόσφατα μία ερώτηση 3 Μαΐου που στην απάντησή μας ε, σε αυτή την ερώτηση λέμε τι γίνεται σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας για την απαγόρευση αυτή. Περιμένουμε τώρα τη συνέχεια της συζήτησης και την έγκριση του σχεδίου ψηφίσματος, αλλά ε, σίγουρα πρέπει να επιβεβαιώσω την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ενδιαφέρον που έχουμε και εμείς, όπως είπαν κύριε Γκροστέτ, κυρία ε, Το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που δρομολόγησε την όλη διαδικασία ε, και την υιοθέτηση αυτού του κανονισμού για τα καλλιντικά και την απαγόρευση των δοκιμών σε ζωή. Είναι δηλαδή πράγματι σκαπανέας πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Προωθήσουμε κατάσταση τροπολογιών 6 Δεκεμβρίου, 11 το πρωί. Στην ΕΜΒΗ θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο του χρόνου. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι... Αχα. Η απαλλαγή του 2016 του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την Κομισιόν Υπηρεσία Περιβάλλοντος ΕΦΣΑ το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών ε, και την Υπηρεσία Χημικών Ουσιών. Μου έδωσαν αυτή την έκθεση οι συντονιστές, οπότε θα σας πω λίγα πράγματα. για την ε, γνωμοδότηση αυτή. Όπως ξέρετε εδώ πέρα κλείνει ο κύκλος του προϋπολογισμού με αυτήν την διαδικασία Κοινοβούλιο και Συμβούλιο εξετάζουν την εφαρμογή του προϋπολογισμού και λογοδοτεί η Κομισιόν και οι άλλοι φορείς όπως και σε προηγούμενα χρόνια θα εκδώσουμε έξι νομοδοτήσεις ε, τις οποίες ανέφερα. Η δουλειά μας ε, στο θέμα της απαλλαγής βασίζεται σε μια έκθεση που κάνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η Κομισιόν και οι υπηρεσίες. Στο σχέδιο γνωμοδότησης εξετάζουμε τα ποσά που είναι διαθέσιμα στην Κομισιόν και στις υπηρεσίες του 2016 για πληρωμές ε, και για πιστώσεις και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Σε γενικές γραμμές τα ποσοστά εκτέλεσης είναι πολύ υψηλά, με κάποιες εξαιρέσεις όπως η Γενική Διεύθυνση Κλίματος για τις πιστώσεις πληρωμών. Επίσης, στο σχέδιο γνωμοδότησης ε, θα βρείτε κάποια σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το έτος 2016, παραδείγματος χάρη, η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου έδειξε μία μικρή μείωση του ποσοστού σφάλματος του τμήματος ε, αγροτική ανάπτυξη, αλία περιβάλλον και κλίμα με 4,9% ενώ το 2015 ήταν 5,3% πλέον. Για το πρόγραμμα LIFE, παραδείγματο χάρη, η Κομισιόν έχει ορίσει ένα σχέδιο δράση μετά τα σχέδια του ελεγκτικού συνεδρίου για να υπάρξει βελτίωση στις καθυστερήσεις πληρωμών και το 2016 το πρόγραμμα έδωσε 315 εκατομμύρια ευρώ για να συγχρηματοδοτηθούν 157 έργα σε 23 κρατη Όσον αφορά τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, τονίζει το βασικό επιστημονικό και τεχνικό έργο τους και κάποιες σημαντικές πρωτοβουλίες όπως αυτές οι οποίες αφορούν την ενίσχυση της διαφανείας. Παραδείγματος χάρη, η υπηρεσία φαρμάκων ξεκίνησε ένα site κλινικών δοκιμών τον Οκτώβριο 2016, δίνοντας έτσι ανοιχτή πρόσβαση σε κλινικές εκθέσεις για τα νέα φάρμακα για ανθρώπινη χρήση που εγκρίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας συνιστώ να τις διαβάσετε. Άρα, με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα και παρά το ότι υπάρχει οπωσδήποτε περιθώριο βελτιώσεων οι έξι εκθέσεις εκφράζουν την ικανοποίησή τους με τη γενικότερη εφαρμογή των τίτλων του προπολογισμού για το περιβάλλον, κλίμα, δημόσια υγεία και ασφάλεια τροφίμων και για τη δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες που είναι υπό την εποπτεία μας και όσον αφορά και την εκτέλεση του προπολογισμού. Οπότε, εκφράζουμε την άποψη ότι μπορεί να δοθεί απαλλαγή στην Κομισιόν σε σχέση με τις δαπάνες ε, στους τομείς αυτούς για το οικονομικό του 2016 και στις πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες που είναι αρμοδιότητός μας. Αυτά εν ολίγης. για την εκτέλεση του προπολογισμού. Θα ήθελα τώρα, αν ενδιαφέρονται και οι ε, σκιοδησηγητές να εκφράσουν την απόψή τους. Θέλει κάποιος να μιλήσει. Η Κάτεμπαχ δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω ποιος θέλει. Μάλιστα, ας ακούσουμε τους κοιόδες συζήτητε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είμαι σκιώδης. Κάποιες φορές σοκάρομαι, τέλος πάντων. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε, κάπως ε, αποσπάστηκε τέλος πάντων. Ε, είμαι σκιώδης από τους Πρασίνους θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχέδια εκθέσεων και για τις απαλλαγές. Ένα σχόλιο μόνο. Λέτε ότι σημειώνετε τις ε, οδηγίες ε, του οργανισμού ε, για τους καταγγέλλοντες από τον EEA. Είναι πολύ καλό που υπάρχει αυτή η διαδικασία, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες εκτελεστικές υπηρεσίες. Επίσης, για την ΕΦΣΑ έχετε ένα σημείο που λέει ότι η αρχή έχει δώσει τα ακατέργαστα ε, στοιχεία που είχε στη διάθεσή της για την ουσία γλυφοσάτη. Αυτό είναι κάπως επίμαχο, πρέπει να πω, διότι ναι μεν έδωσε τα στοιχεία που ήταν ομαδοποιημένα με πίνακες και νούμερα, αλλά τίποτα για τη μεθοδολογία δεν είπαν, τίποτα για τις συζητήσεις δεν είπαν και τίποτα δεν είπαν για τις, ε, τα πορίσματα της μελέτης. Και το σημαντικό είναι ότι τα κάνουν τα δεδομένα όλα αυτά. Αυτή λοιπόν είναι μια σημαντική προσθήκη, πιστεύω που πρέπει να γίνει και αυτός και είναι και ένας λόγος που τώρα πάμε την εύσα στο δικαστήριο τις Βουλευτέ, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια. Και επειδή μιλάτε για τα κατέργαστα αυτά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν, είναι λίγο μονομερές το άρθρο. Γι' αυτό λοιπόν θα καταθέσουμε δύο τροπολίες και έχετε δύο επιλογές. Η μία είναι διαγραφή και τα αφήνουμε ε, το θέμα ε, στην Εύσα... Ε, επειδή το θέμα τώρα έχει, το θέμα τους έχει επιληφθεί το δικαστήριο, άρα δεν λέμε τίποτα. Αν ναι, θα πούμε μια, ε, με μια διατύπωση, και αυτήν την δεύτερη τροπολογία, την όλη ιστορία και να ε, εξηγήσουμε γιατί υπάρχει υπόθεση που θα συζητηθεί στο δικαστήριο, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πληρέστερα. Αυτές ήταν οι δύο τροπολογίες. Ή να μην γίνει καμία συζήτηση στην ε, έκθεση αυτή ή να γίνει πλήρη συζήτηση, να μην νιωθεύσα ότι το Κοινοβούλιο αντιγράφει τα επιχείρηματα και τη ρητορική που χρησιμοποιεί. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλο σκιώδη εδώ. Ποιοι άλλοι βουλευτέ θέλουν το λόγο. Καταρχάς η κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο προλαλή σα, ο Μπασέικ Χάουτ, συνάδελφο. Ιδίω γιατί τι τελευταίε εβδομάδε ε, έχουμε εκφράσει ανησυχίες ε, για την μη δυνατότητα ελέγχου από τον Οργανισμό Χημικών Ουσιών σε ό,τι αφορά τη μη ε, αναγνωρισμένη ε, ως καρκινογόνη ουσία γλυφοζάτη. Και πραγματικά καλό είναι να επαναλάβουμε τις ανησυχίες αυτές. Και ερχόμαστε και ε, στις δύο, στους δύο οργανισμούς, ποια διαδικασία εξολόγησης ακολουθείται, αν είναι διαφανής, τι γίνεται με τους εμπειρογνώμονες και μήπως έχουν και κάποιους δεσμούς με τον κλάδο. Άρα ε, δεν συμφωνώ και εγώ απόλυτα ότι αναπτύσσει τη δημόσια εμπιστοσύνη ε, στο Παγκόσμιο Σύστημα Παραγωγής Τροφίμων, ιδίω λόγω του σκανδάλου τη γλυφοζάτη, λόγω των εγγράφων Μονσάντο και των άλλων αποκαλύψεων, ιδίω στην Guardian και σε άλλε εφημερίδε. Γιατί αυτά όλα δείχνουν τα αντίθετα. Και νομίζω ότι θα πρέπει να τα θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να τα συζητήσουμε εντελεχώ και μετά να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε απαλλαγή ή όχι, ιδίω στους δύο αυτούς οργανισμούς. Κύριε Μπορσάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να πω ότι θα πρέπει να δοθεί απαλλαγή διότι οι πόροι δαπανήθηκαν ε, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Φαρμάκων, η ΕΕ είναι, μάλλον η EMA είναι ένας ε, μια ειδική περίπτωση. Θα πρέπει να μετεγκατασταθεί ο οργανισμός αυτός. Πήρε η απόφαση η Ένωση να πάει στο Άμστερνταμ η έδρα του οργανισμού, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση ο οργανισμός, ιδίως σε ό,τι αφορά ε, το κόστος που σχετίζεται με το Brexit και προσλήψεις ε, που θα χρειαστεί να γίνουν, πρόσθετες προσλήψεις, γιατί πρέπει να αντισταθμιστεί απόλυτα κάποιου προσωπικού, κάποιων μελών προσωπικού. Οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στο Άμστερνταμ, ε, οι περισσότεροι πάλι, κάποιοι όμως όχι. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πλέον κόστος. Επίσης, πρέπει να δοθεί γρήγορα η άδεια για την ε, μεταφορά στο νέο κτίριο. Δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα με την κατάσταση του οργανισμού. Πρέπει και το σύστημα πληροφορικής να συνεχίσει να λειτουργεί για να μπορούν να παρέχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες στους πολίτες. Κυρία Ντορνανό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε ό,τι το γενικό προπολογισμό, Σημειώνω την ανησυχία μου για το ότι η ΔΕΛΤΑ περιβάλλον δεν κατάφερε να συγκρίνει και να παρακολουθεί τι γίνεται ε, με το φόρτο εργασίας. Δείχνουν το 2016 έλεγχοι ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων. Άρα έχουμε ένα ζήτημα. Ποια θα είναι η μελλοντική διαχείριση των εσόδων της Ένωσης που από ό,τι φαίνεται θα μειωθούν με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλη κακή έκπληξη είναι καθυστέρηση στην εφαρμογή των συστάσεων για την ασφάλεια του συστήματος πληροφορίας και την ανταλλαγή των των εκπομπών. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Όπως ξέρετε, αυτό το σύστημα καλύπτει 31 χώρες. 11.000 εγκαταστάσεις, ε, βιομηχανικές μονάδες αλλά και αεροπορικές εταιρείε καλύπτονται από τις ε, συμμετέχουσες χώρες. Φανταστείτε λοιπόν αν το σύστημα αυτό καταρρεύσει. Ξέρουμε ότι οι επιχειρήσεις μας είναι εκτεθειμένες σε έναν παγκόσμιο και συχνά θέμητο ανταγωνισμό σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τι γίνεται τώρα για την ΕΦΣΑ. Θετικό είναι να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη. Να υπάρχει άνοιγμα, να υπάρχει διαφάνεια. Όμως το σκάνδαλο των Monsanto Papers δείχνει ότι στρατηγικοί στόχοι που αναφέρονται στρατηγική 2020 δεν εκπληρώνονται. Δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερο κατόφλι αποδείξεων, αποδεικτικών στοιχείων και να ενισχυθούν οι δυνατότητες επιστημονικής ε, αξιολόγησης. Βλέπουμε να γίνεται μόνο μια αντιγραφή επικόλυση των εγγράφων Μονσάντο. Αυτό δεν δείχνει μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία για την ΕΦΣΑ. Θα καταθέσω για τις διάφορες αυτές απαλλαγές σχετικά τις τροπολογίες που σας εξέθεσα ως προς το περιεχόμενο. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Πολλοί είναι εδώ, δεν ξέρω ποιος θέλει το λόγο. Διαλέξτε. Και να μας λέτε και ποιος είστε κάθε φορά. Okay. Um, for DG Climate Action, thank you, Madam Chair, for giving me the floor. Uh, την DG Climate Action, ευχαριστώ σε το λόγο και, και συνάδελφοι από την μονάδα των χρηματοοικονομικών. Πρώτα πρώτα να δούμε το γιατί δεν προχώρησε η εφαρμογή των εφαρμοστικών μέτρων για το ETS. Εμείς διαχείριζαμε το θέμα και όχι η Γενική για το Περιβάλλον. Υπάρχουν το Μητρό, έχουμε επίσης τις ε, συναλλαγές και αυτά όλα καλύπτονται από μία σύσταση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Οικονομικών Ελέγχων το, και το σύστημα Open. Τα εξή θα πρέπει να γίνει. Υπάρχει αυτός ο χάρτης για την ασφάλεια, θα πρέπει να εφαρμοστεί και το όλον σύστημα θα πρέπει να καλυφθεί από μια πλατφόρμα ασφαλείας στο Λουξεμβούργο. Και μαζί με την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Πόρων προσπαθούμε ούτως ώστε αυτή η υλοποίηση να γίνει το στομότερο δυνατόν. Παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση γιατί πρόκειται για πρωτοπόρα δράση μας ούτως ώστε να έχουν προστασία από τις κυβερνοεπιθέσεις όπως το δεκτατές 2011 Να έχουμε ένα, ένα firewall, ένα σύστημα ασφαλείας όπως θέλετε, πέστε το, ακριβώς όπως έχουν και οι τράπεζες. Οπότε αναβάλαμε την ημερομηνία στόχο και πήγε τώρα το 2018. Τα έλεγε αυτά και η έκθεση πέρσι. Και αυτά γιατί είχαμε υποτιμήσει το πόσο περιπλοκό είναι το θέμα και πόσο χρόνο θέλει για να φτιαχτεί αυτό το σύστημα ασφαλείας. Και μέχρι το τέλος του 2018 ελπίζουμε όλα να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει γίνει όπως τη θέλουμε η εφαρμογή, να κάνουμε την αξιολόγηση κινδύνου, οπότε αν θεωρήσουμε ότι ο κίνδυνος πέραν αυτού είναι αποδεκτός, πλευρά των υπηρεσιών μας θα προχωρήσουμε ακριβώς όπως λέει και η ετήσια έκθεση και θα έρθει η επιφύλαξη που υπάρχει πάντως όλες οι υπηρεσίες συνεργαζόμαστε ούτως ώστε να γίνουν αυτά το συντομότερο ευχαριστούμε πριν ξαναδώσουμε το... Α, θέλει το λόγο πριν προχωρήσουμε κυρία Κάντενμπαχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Εγώ είχα σημειώσει ότι θα ξεκινούσαμε στις 12. Να ήταν λάθος βεβαίω. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την πρόταση αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε την πρότασή σας για τις υπηρεσίες που είναι αρμοδιότητός μας Και βεβαίως θα ήθελα να πω το εξής, ότι όταν αναμένουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένες και με επαρκή προϋπολογισμό αυτές οι εταιρείες. για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ε, απαιτήσεις των Ευρωπαίων. Επίσης σημαντικό είναι να δούμε τις επιδόσεις τους και το νομικό πλαίσιο. Ε, και βεβαίως ε, έχουμε και τις σχετικές συζητήσεις που ανακύπτουν κάθε φορά που μιλάμε για την γλυφοσάτη και το πώς αξιολογούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να αλλάξουμε πιθανώς και το νομικό πλαίσιο. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες έρευνες για το τι γίνεται για τις ε, μελέτες που αναλαμβάνονται σε συνεργασία με την Μονσάντο. Είμαι πεπισμένη ναι. λοιπόν ότι εργάστηκαν πάρα πολύ καλά το 2016, αν δούμε τις λεπτομέρειες ε, του ελεκτικού συνεδρίου και τις παρατηρήσεις που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο που ελήθησαν σοβαρά υπόψη, ειδικά αυτές που αφορούν την διαφάνεια. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να δώσουμε την απαλλαγή. Αυτά σας ευχαριστώ και ελπίζω πάντα τέτοια να είναι η συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεκλέρ λέγομαι τμήματάρχης ε, της αρμόδιας υπηρεσίας. Λοιπόν, καλοδεχούμενη η γνωμοδότηση του ελεγκτικού συνεδρίου για τους λογαριασμούς του 2016. Όπως είπαμε, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα σχέδια δράσης που έχουν αναπτύξει και σαφώς ε, μιλάμε για απαλλαγή για το 2016 και σημειώνουμε όλα τα σχόλια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα κάποιος άλλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξάνδρα Βάκρο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Σε γενικές ε, γραμμές μαζί με τους συναδέλφους από τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος, γιατί όπως ξέρετε από κοινού εφαρμόζουμε το πρόγραμμα LIFE. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την έκθεση αυτή και την απαλλαγή και βεβαίως ε, ακούμε τα πολύ θετικά σχόλια ότι προσπαθούμε δηλαδή να βελτιώσουμε το ποσοστό εφαρμογής. Επίσης προσπαθούμε να μειώσουμε τις καθυστερήσεις της πληρωμές και να δώσουμε τα σχετικά κονδύλια στους δικαιούχους, αλλά στο live και στα άλλα έργα. Και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Επίσης, καλωσορίζουμε τα σχόλιά σας για την απαλλαγή των υπηρεσιών για όλες τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τα σχόλιά σας επίσης για τους πληροφοριοδότες, αλλά και το σχόλιο ότι πρέπει να δούμε σοβαρά το επίπεδο στελέχωσης. Ιδιαιτέρως μιλάμε για την υπηρεσία περιβάλλοντος που εξυπηρετεί και το περιβάλλον και το κλίμα, αλλά και την υπηρεσία χημικών και γνωρίζουμε κάποιες δυσκολίες ε, στελέχωσης αυτών των υπηρεσιών, χωρίς να παραμελούμε το ότι ισχύει αυτό για όλες τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες. Πληροφοριακά, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιολόγηση και θα προκύψουν κάποιες συστάσεις για την στελέχωση. Θα ήθελα μόνο να τονίσω κάτι το οποίο θα θέλαμε να δούμε μαζί σας και την γραμματεία της Επιτροπής για το επίπεδο εφαρμογής ε, των ε, πιστώσεων πληρωμών γιατί θεωρούμε σύμφωνα με τα εσωτερικά μας δεδομένα ότι το επίπεδο είναι ελαφρώς ψηλότερο. Όχι βεβαίως στο 99% της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, αλλά θα θέλαμε ή δυνατόν να διορθωθεί αυτό το λάθος Αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιος άλλος από την Κομισιόν. Όχι. Όχι. Οπότε αν υπάρχει και κάποιος από τις υπηρεσίες αυτές που θέλει τον λόγο για κάποιο θέμα. από την EA, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Θέλω να σας ευχαριστήσω κυρία εισηγήτρια για την άποψή σας, για την γνωμοδότηση και θα διαβιβάσω στην Κοπενχάγη τη θετική σας σύσταση. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος, λέει πρόεδρος? Αν όχι, τότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Πρέπει να πω ότι εκτιμώ όλα τα σχόλια. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές είναι ε, σημαντικές. Περιμένω τους τροπολίες των συναδέλφων. Θέλουμε να έχουμε ε, μια καλή επισκόπηση της κατάστασης και του προπολογισμού για τις έξι αυτές απαλλαγές. Έχουμε ορθισμένα κατάσταση τροπολογιών τη 12η Δεκεμβρίου στις 5 το μεσημέρι. Και 24 και 25 Ιανουαρίου είναι η ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή μας του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Εδώ ολοκληρώνεται η πρωινή συνεδρίαση. Μην ξεχάσετε όμως ότι έχουμε το μεσημέρι ακρόαση και ξεκινάμε στις 2.30 για τις ε, πτώσεις του Brexit. Σας ευχαριστώ.